ακούσουμε τώρα την κυρία Μουσκαρντίνη για μια σύντομη παρουσίαση της έκθεσης ε, για την καταπολέμηση των, ε, του ακροτηριασμού των γυναικείων γενετικών οργάνων που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι ε, πολύ ε, δόκιμο που συμμετέχει στη συζήτηση ο Επίτροπος Μισελ, γιατί ξέρουμε πόσο προσφυλίτου είναι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η παρουσία του Επιτρόπου Μισελ ε, μου δημιουργεί ελπίδες ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσέξει ιδιαίτερα αυτό το πρόβλημα που σήμερα δεν επηρεάζει μόνο τι 28 αφρικανικές χώρες και πολλές ε, χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά ενδιαφέρει και πολλές ευρωπαϊκές χώρες πια. Το πρόβλημα αυτό έχει γίνει φλέγον ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η μαζική μετανάστευση που έλαβε χώρα τα τελευταία χρόνια έφερε την τραγωδία του ακροτηριασμού των γυναικείων γενετικών οργάνων και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεκάδες χιλιάδες κοριτσιών και νεαρών γυναικών κινδυνεύουν καθημερινά να υποστούν μία αποτρόπαια πρακτική που από σωματική τουλάχιστον άποψη δημιουργεί ανεπανόρθωτα αποτελέσματα, ανεπανόρθωτες βλάβες και ταυτόχρονα προκαλεί και ανεπανόρθωτη ψυχική ζημία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που εγκύπτει το θέμα αυτό και μάλιστα μέσω του προγράμματος Δάφνη είχε χρηματοδοτήσει 14 προγράμματα για την καταπολέμηση του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Σήμερα αντιμετωπίζουμε και πάλι όμως το πρόβλημα αυτό, γιατί δυστυχώς αυτό το φαινόμενο του ακροτηριασμού δεν έχει μειωθεί, δεν έχει εξαλειφθεί. Δυστυχώς βρίσκεται ακόμη σε φάση εξάπλωσης. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε το κουράγιο και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε με πιο σωστό τρόπο μία σοβαρή πρόληψη μέσω εκστρατιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο τις ε, γυναίκες μετανάστες αλλά και τους γονείς αυτών των παιδιών. Δεν είναι με μία φιλετική τελετή που δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία μπορεί κανείς ε, να προσβλέπει σε μια καλύτερη κοινωνική ένταξη ή σε μια βελτίωση του μέλλοντος ε, των κορισιών τους για παράδειγμα μια, ένα κορίτσι που πηγαίνει σε γαλλικό, βελγικό, ιταλικό σχολείο και που μετά από συναναστροφή με τις ε, συνομήλικές της ε, ξεφεύγει από την πραγματικότητα και υφίσταται μια τραγωδία που την ε, σφραγίζει για την υπόλοιπη ζωή της και σωματικά και ψυχικά η κοπέλα αυτή δεν θα ακροτηριαστεί μόνο σωματικά, αλλά θα βρίσκεται πια σε αδυναμία να συναναστραφεί επίσης όρις ε, τους ε, συνομιλίκους της. Θα είναι πια διαφορετική και εμείς δεν θέλουμε διαφορετικούς ανθρώπους στην κοινωνία μας. Θέλουμε ε, ανθρώπους που πέραν της θρησκευτικής τους ή της πολιτικής τους ιδεολογίας ή της γεωγραφικής προέλευσης να συμβάλλουν όλοι μαζί σε μια καλύτερη Ευρώπη, σε μια καλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και ευχαριστώ όλους τους υπαλλήλους επιτροπείς που με βοήθησαν να συντάξω την έκθεση. Θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία εναρμόνιση των κρατικών νομοθεσιών προκειμένου να στοιχευτηθεί ως έγκλημα ο ακροτηριασμός των γυναικείων γενετικών οργάνων. Δεν θέλουμε να, να προταθούν εναλλακτικές λύσεις όπως αυτή η εναλλακτική ένεση. Δεν θέλουμε τέτοιες ε, τελετές μοίησης, θέλουμε πραγματική ένταξη των μεταναστών στις κοινωνίες μας. Θέλουμε οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις να μπορέσουν να εργαστούν, θέλουμε μια πρόληψη στη συνεργασία με τις γυναικείες οργανώσεις ε, των μεταναστών. Θέλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αποφευθεί αυτός ο ακροτηριασμός των κοριτσιών που τις φέρνει σε ένα φαύλο κύκλο περιθωριοποίησης και απομόνωσης. Ελπίζω οι συνάδελφοι να εξέτασαν αυτό το θέμα και να στάθμισαν τις ολέθρες συνέπειες του και νομίζω ότι μπορούμε να απευθύνουμε μια έκκληση προς μια ισχυρότερη Ευρώπη για συνεργασία των θεσμικών της οργάνων προκειμένου να αποτεχθεί αυτό το ε, αποτρόπαιο έγκλημα που καταστρατηγεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό θα πρέπει να είναι ο κοινό μας στόχος. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ο κύριος Μισελ έχει το λόγο. <clears throat> Θα ευχαριστήσω όχι τη συναδέλφου μου αλλά και προσωπικά την κυρία Μουσκαρδίν γιατί εδώ μιλάμε για ένα πραγματικό δράμα και ένα σκάνδαλο συγχρόνως. Θέλω να ευχαριστήσω κυρία Μουσκαρδίν για τη θαυμασία εκθεσή της και για τη σημασία, θα εξάρτητα τη σημασία του αγώνα κατά του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν το έχει καταγγείλει τόσο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις τρίτες χώρες ότι αυτό είναι μια πρακτική παραδοσιακή απαράδεκτη η οποία πλήττει την σωματική ακαιρεότητα των γυναικών και των κοριτσιών όχι μόνο τη σωματική του ακαιρεότητα και την ψυχική του ακαιρεότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο από τι τρίτε χώρε αλλά και από τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση με στεναρά μέτρα, ακόμα πιο στεναρά μέτρα γιατί εξακολουθεί όσο απίστευτο και να φαίνεται να εξακολουθεί να ισχύει αυτή η πρακτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν αυτή η πρακτική να σταματήσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω από αυτήν. Μέσα στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου που έχουμε με τι τρίτε χώρε θα πρέπει να υπογραμμίζεται το θέμα αυτό και θα πρέπει να γίνεται κατανοητή η θέση μα αυτή. Βγαίνω λιγάκι από το κείμενό μου και θέλω να τονίσω ότι σε κάθε πολιτικό διάλογο που έχουμε με τι αναπτύσσόμενε χώρε ιδίω, κάθε φορά στην μέση διάταξη είναι αυτό το θέμα. Πολύ πρόσφατα, παραδείγματο χάρη, ο πρόεδρος Καμπαρέ του Μπουρκίνα Φάσου με πήρε στο τηλέφωνο λέγοντα ότι είναι έτοιμοι να περάσουν νομοθεσία η οποία θα απαγορεύσει αυτή την πρακτική στον Μπουρκίνα Φάσο, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχουν ορισμένες φυλές, ορισμένες φατρίες οι οποίες εφαρμόσουν αυτές τις πρακτικές και είναι ένα ευαίσθητο θέμα, αλλά υπήρχε πολιτική θέληση να εφαρμοστεί από τον Μπουρκίνο Φάσο αυτό. Η Κομισιόν έχει δώσει κοινοτικά κονδύλια για να υποστηρίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρίτε χώρες την αντιμετώπιση αυτών των ακροτηριασμών και επίσης να βοηθηθούν τα θύματα και τα νέα κορίτσια τα οποία κινδυνεύουν με, από αυτή την πρακτική. Έχουμε το πρόγραμμα Δάφνη 3 το οποίο υποστηρίζει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις δημόσιες και τοπικές ή περιφερειακές αρχές των τρίτων χωρών για τον αγώνα κατά του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και έχετε πει και εσείς ότι η Δάφνη έχει χρηματοδοτήσει 14 ειδικά προγράμματα σε ύψος 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο στόχος είναι η κατάρτιση, η υποστήριξη, η δράση ευαισθητοποίησης, η συλλογή στατιστικών πληροφοριών, η ανάπτυξη εργαλείων και η δημιουργία βελτίστων πρακτικών στον τομέα αυτό, και η απαραίτητη υπαρχή πληροφοριών στους λήπτες αποφάσεων. Φυσικά θέλουμε να διατηρήσουμε την υποστήριξή μας στις δράσεις αυτές και να εξακολουθήσουμε να έχουμε επιτάπητο στο θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια της πρόληψης της βίας και στην, στα πλαίσια της αρρωγής των θυμάτων αλλά και σε ό,τι αφορά την ε, μετανάστευση, την παροχή ασύλου και την ποινική δικαιοσύνη. Αντιμετωπίζουμε από όλες αυτές τις οπτικές γωνίες το πρόβλημα αυτό και εγώ πραγματικά σοκάρομαι βαθύτατα, πρέπει να το πω, για την δηλία ορισμένων κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων πολιτικών που θεωρούν ότι αυτό είναι ένα πολιτιστικό ζήτημα και επομένω δεν μπορούμε να επέμβουμε. Όχι. Αυτοί οι οποίοι έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τύχουν σεβασμού των κανόνων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να έχουμε δικαιοσύνη, δεν μπορούμε να έχουμε δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Δεν μπορούμε να έχουμε αρχές δύο ταχυτήτων. Αυτό θίγει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ έχω συμβάλει σε αυτή τη συζήτηση στο παρελθόν και πραγματικά είναι ένα σκάνδαλο το γεγονός ότι ορισμένοι με το πρόσχημα της διαφορετικής πολιτισμικότητας των μεταναστών αρνούνται να ποινικοποιήσουν τέτοιες πρακτικές. Τουλάχιστον θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πρακτική μέσα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να παρακάμψουμε την ανάγκη να πούμε ότι οι κανόνες μας, τα συντάγματά μας, οι ανθρώπινες αρχές μας εμποδίσουν μια τέτοια πρακτική και είναι παράνομη εκτός νόμου και αξιόπινη αυτή η πράξη. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορώ να πω ότι σίγουρα συμμερίζομαι την αγανάκτησή σας για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά την βοήθειά της προς τρίτες χώρες, η Κομισιόν έχει αναπτύξει πολιτικές εναντίον του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων γιατί αυτό είναι και θέμα χειραφέτησης των γυναικών, δικαιωμάτων ανθρωπίνων των παιδιών και τμήμα του πολιτικού και στρατηγικού διαλόγου που κάνει με τις εταίρες κυβέρνηση, κυβερνήσεις. Υποστηρίζει επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση όλες τις δράσεις υποστήριξης ενώπιον των κυβερνήσεων των εμπλεκομένων χωρών και όλες τις προσπάθειες για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την απαγόρευση όλων των πρακτικών που φύγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης θέλουν να, θέλουν να αυξήσει τις δράσεις των πολιτικών υπευθύνων και τις δράσεις του πληθυσμού και όλων των εμπλεκομένων. Τα πολυετή προγράμματά μας λοιπόν καλύπτουν μια σειρά δράσεων που έχουν σαν στόχο να αναπτύξουμε ένα χώρο δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας μέχρι το 2010 και μέσα στα πλαίσια αυτά θα παρουσιάσουμε το νέο πρόγραμμα της Στοχόλμης 2010-2014 την άνοιξη του 2009 και το πρόγραμμα αυτό θα <clears throat> δώσει μεγάλη έμφαση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία των δικαιωμάτων των ε, θυμάτων, μεταξύ των οποίων και των δικαιωμάτων των γυναικών. Η Κομισιόν δεν έχει ακόμα αναπτύξει μια ειδική στρατηγική για τον αγώνα κατά τον ακροτηριασμό των γυναικείων οργάνων, αλλά είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την απαραίτητη προσπάθεια σε δράση προ την κατεύθυνση αυτή και θέλουμε να συνεχίσουμε να θέτουμε το θέμα αυτό στι εσωτερικέ αλλά και εξωτερικέ πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Συνεχίζουμε τώρα με την τελευταία έκθεση στην ημερήσια διάταξη του κυρίου Γκρασαμόρα για την πολυγλωσία. Ένα κοινό εγχείρημα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ανακοίνωση της Κομισιόν με τίτλο